λόγο. Η θέση της ε, Κομισιόν για κάθε μία από τι τροπολογίε είναι διαθέσιμη σε εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο και περνάμε στο, επόμενο σημείο η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και αυξημένε ελεκτρικές εξουσίε τη Ευρώπη μέσω τη Eurostat. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Ότμαρ Κάρας για δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι ρεν, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή συζήτηση είναι σημαντικό πολιτικό μήνυμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλει να εκπέμψει αυτούς τους καιρούς. Είναι επίσης και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας με την προφορική αυτή ερώτηση μεσούς της διαδικασίας της ε, αναδιάθρωσης της Eurostat και ε, την γνωμοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα ίδιο ψήφισμα δείχνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια ευρύτατη ανεξάρτητη λειτουργία της Eurostat και τη χρειάζεται, όχι μόνο ότι θέλει. Είναι η πρώτη άμεση νομοθετική επίπτωση των καταστάσεων με την Ελλάδα. Το Συμβούλιο ε, το 2005 αρνήθηκε ε, και το, ε, την πρόταση του κ. Αλμούνια και ε, δεν θέλησε να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε εδώ και καιρό να τα είχαμε κάνει αυτά. Οφείλαμε να τα είχαμε κάνει, όχι μόνο το επιθυμούσαμε. Αλλά και την Κομισιόν και το Συμβούλιο θέλω να προειδοποιήσω και να πω ότι υπάρχει πολιτική βούληση να έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε έτσι ώστε το ευρώ να μην παραμείνει μόνο στην νομισματική ένωση, αλλά να έχει και ένα σκέλος οικονομικής ένωσης και να μπορεί να πατάει και στα δύο αυτά πόδια. Και παρακαλώ το Συμβούλιο να μην αποτρέπει, να μην χρονοτριβεί, να μην παρεμποδίζει, αλλά να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα πράξει όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι, επίσης θέλουμε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν έρευνες για παραλήψεις, ατασταλίε τα τελευταία χρόνια στη Eurostat στα κράτη-μέλη. Γιατί μόνο όταν έχουμε μια σαφή ανάλυση μπορούμε να γνωρίζουμε και τι διορθώσεις χρειάζονται και τι συμπληρώσεις χρειάζονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θέλει. Ανεξαρτησία, συγκρισιμότητα των στοιχείων, γι' αυτό ελάχιστες προδιαγραφές για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και για τη θεσμική συγκρότηση ε, των ε, στατιστικών αρχών και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλουμε τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα και να μπορούν να ελέγχονται ανα πάσα στιγμή χωρίς προέγκριση. Επίσης θέλουμε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία και σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο κοινωνικών ασφαλίσεων και ε, για αρμονική συνεργασία και συντονισμό. Επίσης επιθυμούμε πριν ολοκληρώσουμε τη ε, δραστηριότητά μας, αν ε, όλα αυτά που κάνετε είναι επαρκή, δεν θέλουμε τα ελάχιστα θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα προς την ανεξαρτησία και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Eurostat. Κάρας, la parola Presidente Sharon uh, thank you. The Economic and Monetary Affairs Committee is... Η Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, είναι συνεπής και ενωμένη και εμένουμε το ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η Eurostat και ότι Όπω λέμε εδώ για πολύ καιρό, ότι θα πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα τα αστικά δεδομένα και όπω το είπε ο κύριο ε, Κάρα, πάντα ισχύουν αυτά. Το 2005 ε, αυτά που αποφάσισε το Συμβούλιο ήταν για, για, για ντροπή, ιδίω όσον αφορά το κυρίαρχο χρέο και όσον αφορά το ε, σύμφωνο σταθερότητα. Γιατί εάν κανένα δεν κάτσει και να μελετήσει την ιστορία, να λάβει το ιστορικό πλαίσιο, είναι δύσκολο κανεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη, ιδίω με τη σημερινή συγκυρία που το πράγμα είναι τόσο δύσκολο, γιατί είδατε πόσα χρήματα εκταμείευσαν ε, τα, τα, τα, τα, κράτη και δεν ήταν ε, αρκετές οι αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ. Όντω θα πρέπει σύντομα να έχουμε αυξημένε ελληνικέ ομάδε από την Eurostat και το σούτο μάλλον μια που σήμερα χρειάζεται αυτό γιατί αυτό θα είναι το κλειδί ούτω ώστε η οικονομική υποπτία να είναι αποτελεσματική και γι' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καινούργιο ε, εργαλείο ε, το οποίο να κάνει τι υποσχέσει πράξη. Θέλουμε επομένω να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, θέλουμε αυτά να γίνονται με σωστό timing και επίση θέλουμε να μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε ε, μια συνεισφορά στους εθνικούς λογαριασμούς και άρα γι' αυτό θα πρέπει να έχει ε, τις αρμοδιότητες που πρέπει η Eurostat. Τώρα, έχει τάξει κάποιες όρους και προϋποθέσεις στο ΕΚΟΦΗΝ. έτσι υπονομεύει το να μπορεί έγκαιρα να παρέμβει και να ελέγξει ε, η Eurostat. Εμείς θέλουμε γύρω στα να έχει τις σχετικές αρμοδιότητες χωρίς καμία προϋπόθεση και περιορισμό και να μπορεί να κάνει αυτές τις μεθοδολογικέ επισκέψεις. Βεβαίω και θα πρέπει να στοχοθετήσουμε τους πόρους μας εκεί που χρειάζεται, αλλά η έρευνα θα πρέπει να γίνεται εκεί που χρειάζεται όταν γεννηθεί υποψία και όχι εκ των υστέρων. Τέλος, πότε θα μάθουμε ότι πρέπει να συγκρίνουμε συγκρίσιμα και ότι θα πρέπει να υπάρχει προτυποποίηση και διαφάνεια στους ελέγχους, ούτως ώστε να μπορούμε ό,τι καινοτό, καινοτόμες ενέργειες και πονηρές υπάρχουν, μπορούμε να τις πιάσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα το λόγο έχει όλοι Ρένο, Επίτροπος. President, uh, honorable members, uh, let me first uh, thank you Uh, Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάρας ε, και αλλούς ε, για το ότι έθιξαν αυτό το τόσο σημαντικό θέμα όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων της Eurostat. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υποστήριξη που προσφέρατε στην πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλου για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να υπογραμμίσω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την πρώτη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής Μπαρόζο. Και ελπίζω αυτή η πρόταση να εγκριθεί σύντομα και κατόπιν την πρόταση αυτή θα τη συμπεριλάβουμε στο οπλοστάσιό μας. Βεβαίως την είχαμε χρειαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως είπε και η κυρία Πόουλς. Το 2005 έγινε η αρχική πρόταση, τότε όμως απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη. Βέβαια, οι καιροί έχουν αλλάξει και τώρα επιτύχαμε ευρεία υποστήριξη στο Συμβούλιο. Όσον αφορά λοιπόν στην πρόταση αυτή, η γενική προσέγγιση ε, συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στις 8 Ιουνίου την περασμένη εβδομάδα και το γεγονός αυτό υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ποιοτικά δεδομένα όσον αφορά κυβερνητικά ελλείμματα. Επίσης αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κομισιόν και της Eurostat για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ο κανονισμός ε, αφορά στον ε, βασικό στόχο της ε, πρότασης που κατέθεσε η Κομισιόν, δηλαδή να εκχωρηθούν περισσότερες ελεγκτικές αρμοδιότητες στη Eurostat οποτεδήποτε εμφανίζεται πρόβλημα σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων. Κατόπιν τούτου η Κομισιόν δέχεται το συμβιβαστικό κείμενο. Η Κομισιόν προτίθεται να λάβει και άλλα μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στοιχείων. Ε, θα υπάρξει άμεση ενίσχυση των πόρων που διατίθενται για το προσωπικό. Κυρίως ε, θα γίνει και εσωτερική ανακατάταξη στο προσωπικό. Ε, τα κράτη-μέλη θα δέχονται πολύ πιο συχνά επισκέψεις από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα η Κομισιόν θα διασφαλίσει την ακαιρεότητα των πηγών από τις οποίες προέρχονται τα στοιχεία, όπως προβλέπει ο κανονισμός, και αν προκύψει μια κατεξαίρεση περίπτωση για ιδιαίτερο κίνδυνο, οι προβλήματα όσον αφορά ε, στην ποιότητα των στοιχείων, τότε η Eurostat θα χρησιμοποιήσει όλες τις ε, αρμοδιότητες που έχει στη διάθεσή της με βάση τον νέο κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των ε, ελεγκτικών αρμοδιοτήτων. Πριν λοιπόν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λιγάκι στην Ελλάδα. Δράτω με αυτή τη ευκαιρία και θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό του χρόνου σα να το χρησιμοποιήσω για αυτό το θέμα. Όπω πολύ καλά γνωρίζετε, η Κομισιόν έχει προβεί σε ενδελεχή έλεγχο των στατιστικών δεδομένων τη Ελλάδα ε, εδώ και τα τελευταία χρόνια. Ο τροποποιημένος κανονισμός ε, προβλέπει να αμβλύνει τον κίνδυνο απάτης ή χειραγώγησης στατιστικών στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανομαλίας, αριθμίας. Εχθές είχαμε μία νέα εξέλιξη όσον αφορά στην Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι ο οίκος Μούντις αποφάσισε να υποβαθμίσει εχθές ένα ελληνικό ομόλογο και αυτό το συζήτησα και με τον συνάδελφό μου κύριο Μισελ Μπαρνιέ και με τον πρόεδρο της Κομισιόν. Και πρέπει να πω ότι η απόφαση ο χρονισμός, το timing που η Moody's, ο Moody's ε, έλαβε ε, αυτή την απόφαση είναι λανθασμένος γιατί έρχεται ακριβώς μετά τη συμφωνία που συνήψε η Ελλάδα με την Επιτροπή, ε, το Διεθνές Δομιλωτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή και την Τράπεζα για, την, για το νέο πρόγραμμα που θα εφαρμόσει. Οι αποφάσεις που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση καταδεικνύουν τη στράτευσή της να τροποποιήσουν το στατιστικό σύστημα της χώρας, να εξηγιάνουν τα οικονομικά και να δρομολογήσουν μία βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν η απόφαση του οίκου είναι ασυνεπής ε, με τις ε, ελληνικές αποφάσεις ε, και με τα spread που αφορούν στην Ελλάδα που μειώθηκαν σημαντικά από τότε που έχει δρομολογηθεί το νέο πρόγραμμα. Άρα δηλαδή τίθεται πάλι το θέμα του ρόλου των οίκων αξιολόγησης ε, όσον αφορά ε, στις αξιολογήσεις τους. Τα θέματα λοιπόν αυτά θα ληφθούν υπόψη στις ε, απόψεις της Κομισιόν στο μέλλον σχετικά με το πώς θα αξιολογούν τους οίκους αυτούς. Κατά τους επόμενους μήνες η Κομισιόν θα ασχοληθεί με το θέμα του ανταγωνισμού ανταγωνισμού επίσης θα ασχοληθεί με τη διαφάνεια που είναι απαραίτητη σχετικά με το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Γιατί αυτή τη στιγμή ισχύει η αρχή ότι ο πληρώνων επηρεάζει και εκδίδει και τα δεδομένα. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν ότι είναι καθοριστική σημασία να έχουμε ακριβή και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα για τους εθνικούς λογαριασμούς. Γιατί αυτό αποτελεί έναν από τους πυλώνες της εύρυθμα λειτουργούσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο κύριος Κάρας. Η ε, τροπολογία για τις εξουσίες της Eurostat ε, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ε, επιβολής της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, κάτι που είναι ένας απαραίτητος στόχος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει ο κύριος Έντουαρτ Σικλούνα για δύο λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφερε κάποιε νομοθετικέ προτάσει για να τονώσει το καθώς που διέπει την Eurostat, Ακριβώ όπω εξετάστηκε και από την Οικονομική Επιτροπή, γιατί τα στατιστικά είναι το κλειδί για έξω από την κρίση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πώ να πρέπει να δώσουμε τι ευρύτερε αρμοδιότητε, τόσο ώστε να μπορεί να κάνει τι επιθεωρήσει στα κράτη-μέλη. Οι Eurostat όμω αυτέ δεν θα πρέπει δεν είναι μόνο οι συναντήσεις με τους επισήμους, ε, στα Υπουργεία και ε, με τους ελεγκτικούς εθνικούς φορείς. Θα πρέπει νομίζω οι έλεγχοι να μπορούν να καλύψουν ό,τι θεωρείται σημαντικό, δηλαδή με οικονομολόγους, με συνδικαλιστές, ε, με πανεπιστημιακούς, γιατί θεωρούμε ότι αυτό τον τρόπο να προχωρήσουμε είναι αυτονόητο. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό λογιστικό σύστημα το οποίο να το χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη, το οποίο να βασίζεται σε κάποια ε, τυποποιημένα κριτήρια και θα πρέπει να συμφωνηθεί από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και αυτό να μην αφορά μόνο τους, ε, τις οικονομικές εκθέσεις αυτές τις οποίες χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται ως μέθοδος και στο ιστορικό των κρατών μελών, διότι έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που ε, ξεκίνησε η Ευρωζώνη, από τότε που αποκτήσαμε το ευρώ και τώρα ε, βρήκαμε αυτά τα, μεγάλα κενά στο σύστημα το οποίο είναι τόσο ζημιογόνα. Θα πρέπει επομένω να παραδεχτούμε ότι ε, είναι ηρωνία το ότι ήταν τόσο πετυχημένο το ευρώ που αγνοήσαμε αυτά τα κενά στο σύστημα. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον οι αγορέ θα πρέπει να εμπιστεύονται τι στατιστικές και τις προβλέψεις, τα προγνωστικά για τις αγορές. Άρα θα πρέπει να άρουμε αυτά τα κενά στο σύστημα, επομένως θα πρέπει να συνεργαστεί στενά η Κομισιόν με Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και αυτά τα προβλήματα να επιληθούν κατεπηγόντως. Ευχαριστούμε κύριε Σύγκλωνο Πρόεδρος και τώρα. Ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Σίλβη Γκουλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Η σημερινή κρίση της Ευρωζώνης δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο ε, οφείλεται τι κοινέ αριστικές. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι συνέπειε και οικονομικές, αλλά και όσον αφορά την έλλειψη αξιοπιστίας, απόλυτη αξιοπιστίας τη Ένωση, Ένωσης. Γι' αυτό και κατά γνώμη είναι σοβαρό το πρόβλημα, το πώς λειτουργεί σήμερα η Ένωση. Δίνουν υποσχέσει στον κόσμο οι κυβερνήσεις, και λένε ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά τον έλεγχο των δεσμεύσεων των υποσχέσεων και ότι θα μελετήσουμε τα κριτήρια 3,0 δηλαδή. Οπότε βλέπετε τι γίνεται, ότι θα πρέπει να αποκτήσει τα εργαλεία να κάνει τη δουλειά της η Eurostat και όλα αυτά τα οποία έχουν αδυνατήσει τη θέση της, τη θέση της Κομισιόν είναι κάτι κακό για όλους. Άρα θα πρέπει να προωθηθεί αυτό το κείμενο το οποίο ζητεί. Η Eurostat να έχει ευξημένε ελεγκτικές αρμοδιότητες και επίσης να αναδειχθούν κάποια κοινά πρότυπα και επομένως θα πρέπει να υπάρχει τέτοια αυστηρότητα όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, η ιδάλλως θα υπάρχει αποπροσανατολισμός και τελικά αυτό που θα αμαυρωθεί θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Γκουλάρ. Ένα λεπτό, κύριος Όμπερμαϊα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Eurostat δεν αντιμετωπίζει σωστά πραγματικά το πρόβλημα. Δεν θα πρέπει ποτέ ξανά ε, μια χώρα να μπορεί να ε, κάνει τρίκ ε, και να παρουσιάζει πλαστά στοιχεία του προπολογισμού και να ζει πάνω από τις δυνατότητες για πολλά χρόνια εις βάρος άλλων χωρών. Αλλά δεν θα πρέπει να πάρει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αφορμή την Ελλάδα για να ε, μας αφαιρέσει όλες τις αρμοδιότητες στις λειτουργίες μας. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση και η κοινωνική και η οικονομική από χώρα σε χώρα και η Eurostat θα πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό. Ας πούμε ένας άναργος στο Λονδίνο είναι κάτι άλλο από ένα άνεργο στο Παρίσι, διότι τα κριτήρια είναι τελείως διαφορετικά. Ε, και ακόμα πιο κατάφορες είναι οι διαφορές ε, κοινωνικο-οικονομικών πραγματικότητων ε, των χωρών που έχουν σκληρό νόμισμα με τις χώρες που δεν έχουν σκληρό νόμισμα. Αυτός ο μύθος της συγκρισιμότητας δεν θα πρέπει να παραμείνει, θα πρέπει να σπάσει και να τα ξανασκεφτούμε αυτά πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ποδηματά, παρακαλώ. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για το σχόλιο που κάνατε πριν από λίγο σχετικά με την ε, χθεσινή ευνηδιαστική και ανετιολόγητη απόφαση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης moody's να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδα, απόφαση που χαρακτηρίσατε ασυνεπή και λανθασμένη επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ορθότητα τη απόφασή μα να προχωρήσουμε σε μια ριζική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργία των οίκων αυτών στην ευρωπαϊκή επικράτεια και να εξετάσουμε σοβαρά την πιθανότητα δημιουργία ενός δημόσιου ευρωπαϊκού οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης. σε ό,τι αφορά στη σημερινή συζήτηση όπως και στην πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο γνωρίζουμε όλοι ότι έρχεται σε συνέχεια της λεγόμενης ελληνικής υπόθεσης ό,τι αφορά την παραποίηση των στατιστικών δεδομένων και ω ελληνίδα Ευρωβουλευτή είναι προφανές ότι δεν αισθάνομαι ευτυχής που η ελλάδα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα προς αποφυγή για μια τέτοια συζήτηση. θέλω όμως να υπενθυμίσω το κάνατε κι εσείς κύριε επίτροπε ότι η ελλάδα η σημερινή ελληνική κυβέρνηση ήταν αυτή που πρώτη αναγνώρισε το πρόβλημα και πήρε αμέσω ρηξικέλευτε αποφάσει για την αντιμετώπιση του πρώτα απ' όλα με τη μετατροπή της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας σε πλήρως ανεξάρτητη αρχή εποπτευόμενη από τη βουλή και δεύτερον δρομολογώντας τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες όσων έχουν εμπλακεί σε αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται με καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς υπήρξαν επαρκή στοιχεία που θα έπρεπε να μας έχουν κινητοποιήσει ήδη από το. 2005. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Στόγιανοφ. Εγώ θα ήθελα να προσανατολίσω τη συζήτηση σε μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Επίτροπος την περασμένη εβδομάδα εξήγηλε ειδικό έλεγχο για τη Eurostat σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρίας. Δυστυχώς, ο κύριος Ρεν δεν ανέφερε γιατί χρειαζόμαστε τέτοιο έλεγχο για τη Βουλγαρία. Και θα ήθελα να του κάνω συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια ήταν τα κριτήρια που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση την Eurostat. Γιατί τη θεωρείτε χώρα μη αξιόπιστη τη Βουλγαρία. Τη Βουλγαρία που είναι η πιο σταθερή χώρα των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τι από αδράνεια, έτσι από κεκτημένη ταχύτητα. Ε, μετά τη διεύρυνση στραφήκατε προς τη Βουλγαρία. Σήμερα συζητούμε για την Ελλάδα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. αν είναι αυτά τα κριτήριά σας και τώρα έρχεστε να κατηγορήσετε τη Βουλγαρία, αυτό μπορεί αυτόματα να επηρεάσει και την αξιολόγηση των οίκων προς τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλά είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επικρατήσει σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα ευκολότερα αλλά και τα πιο σημαντικά μέτρα, πιο σημαντικό, είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Είναι λοιπόν εύκολο να βελτιωθεί η κατάσταση, σημαντικά μάλιστα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να χαιρετήσω τις θετικές κινήσεις τόσο από την Κομισιόν όσο και από το Συμβούλιο προς αυτή η κατεύθυνση. Εγώ προτείνω ταχύτατα να εγκρίνουμε τη δέσμη μέτρων που θα βελτιώσουν την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος αλλά και οι αρμοδιότητες της Eurostat. Η Eurostat ε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, όμως ε, οι αποφάσεις ε, και η ιεράρχηση ε, θα πρέπει να είναι σαφέστερη. Η Eurostat πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχει στον έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλονται και πρέπει η Eurostat ε, να μπορεί να διεξάγει ελέγχους ε, οποτεδήποτε κρίνει ότι η ποιότητα είναι ανεπαρκής. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να αυξηθούν οι πόροι. Η υψηλή ποιότητα ε, ε, απαιτεί και υψηλότερες επενδύσεις. Πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα για τη Eurostat, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά της και το προπολογισμό να επιτρέπει τέτοιο περιθώριο για τη βελτίωση της ποιότητας. Εγώ ανησυχώ γιατί σήμερα τα στατιστικά στοιχεία δεν αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα και ελπίζω στο μέλλον να υπάρχει αύξηση των πόρων προς επίτευξη του στόχου αυτού. Τώρα πάμε στο Catch the Eye και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μόλσεν. Γνωρίζουμε όλοι μας ε, ότι όσον αφορά τον κανονισμό για την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων ε, αυτή η πρόταση ε, δυστυχώς δεν καλύπτει τα προβλήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, όμως είναι ένα απαραίτητο μέτρο. Γιατί ε, μόνο εφόσον υπάρχουν σωστά μέτρα μπορούμε να λάβουμε, μάλλον σωστά στοιχεία μπορούμε να λάβουμε και σωστά μέτρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου έτσι ώστε τα στοιχεία που καταθέτουν οι κυβερνήσεις να μπορούν να ελεγχθούν έγκυρα. Ε, δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό που έγινε με την Ελλάδα. Δηλαδή εκ των υστέρων ε, με βάση παραποιημένα στοιχεία να έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις και πρέπει να τιμωρηθούν τα κράτη εκείνα τα οποία δόλια υποβάλλουν παραποιημένα στοιχεία. Η ε, προώθηση, η προαγωγή της Eurostat ως ανεξάρτητο οργανισμό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνουμε στην ε, δημοσιονομική, ε, ε, στη δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών. Απλά θέλουμε να βελτιώσουμε τη Eurostat. Κυρία Γιακονσάρη. Arvoisa Minusta komissiota on syytä kiittää siitä, että... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια που πραγματικά έχει επιτευχθεί ταχεία πρόοδος. Πριν από λίγους μήνες μόλις λέγαμε ότι εάν υπάρξει επέμβαση στα στατιστικά δεδομένα ενός κράτους αυτό σημαίνει παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα επομένως έγιναν βήματα πρόοδου. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αλλίωση των στατικών δεδομένων εκ μέρου μιας χώρας. Όταν γίνεται αυτό, αμαυρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι φταίνε οι Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν λάβει αποφάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους πολίτες ούτως ώστε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Δεν ήταν Ο κύριος Ρέν τώρα. Παρακαλώ όμως να μην κάνετε τόση φασαρία. Uh, Αγαπητά μέλη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας ευχαριστήσω για αυτή την ουσιαστική συζήτηση που προέκυψε και για την υποστήριξή σας ε, στην πρότασή μας που είναι να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες της Eurostat. Και πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Γιακονσάρη. Δηλαδή πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική πολιτιστική αλλαγή όσον αφορά την ε, προσέγγιση απέναντι στις οικονομικές πολιτικές στην Ευρώπη. Αυτό αφορά τους τελευταίους μήνες. Η έγκριση λοιπόν αυτής της πρότασης πράγματι θα είναι ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθειά μας ενίσχυσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αναφέρθηκαν διάφορες παρατηρήσεις σε, σε σχέση με την Ελλάδα αλλά και τη Βουλγαρία. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω κάτι και να τοποθετηθώ σε ορισμένα από αυτά που ελέγχθησαν σήμερα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε αυτήν την ιστορία, ολόκληρη αυτή την ιστορία και θέλω όμως να πω ότι δεν είναι σωστό να συνεχίσουμε την ίδια μυθοπλασία γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και εφαρμόζει ένα σωστό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα χρήζει υποστήριξης και όχι κριτικής. Όσον αφορά τις ε, στατιστικές ε, μεταρρυθμίσεις συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές. Έχουμε επισκεφθεί επανειλημμένα την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης και μόλις πρόσφατα συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού ε, συστήματος στατιστικών δεδομένων. Όσον αφορά τώρα στη Βουλγαρία, οι ανησυχίες μας έχουν σχέση κατά κύριο λόγο με δύο θέματα δύο θέματα που αφορούν στις ε, δημοσιονομικές προβλέψεις. Εγώ εμπιστεύομαι τους ευρωβουλευτές από τη Βουλγαρία. Τους άκουσα πολύ προσεκτικά ε, στις τοποθετήσεις τους ε, σε αυτά που είπα εγώ ότι υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα στη Βουλγαρία και υπάρχουν και στατιστικά προβλήματα. Καταρχήν, να σας πω ότι η Επιτροπή μόλις πρόσφατα ενημερώθηκε από τη Βουλγαρία για τις ε, αλλαγές ε, που θα υπάρξουν στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και στην παραβίαση των υποχρεώσεων της Βουλγαρίας που απορρέουν από την υπογραφή της συνθήκης ένταξής της. Δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε γιατί η Βουλγαρία αναθεώρησε τον προπολογισμό της για το 2010 από έναν ισοσκελισμένο προπολογισμό πέρασε σε έλλειμμα 3,8%. Αυτό το μάθαμε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ε, παρότι το μακροοικονομικό σκηνικό παραμένει αναλύωτο. Κατόπιν τούτου, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δημοσιονομικές προβλέψεις της ε, Βουλγαρίας για φέτος. Η Eurostat θα επισκεφθεί τη Βουλγαρία κατά το δεύτερο ήμιση αυτού του έτους και κατά διάρκεια αυτής θα εξεταστούν οι διαφορές, οι τροποποιήσεις ε, σχετικά με τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Η Eurostat θα εστιάσει την προσοχή της ε, σε ενδυνάμει κινδύνους, στο ότι μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις όσον αφορά τη διαδικασία σε σχέση με το 2009 και σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Βουλγαρία. Ε, προσέχω πάρα πολύ και ε, θέλω να πιστήσω και τη δική σας την προσοχή ότι αυτό το θέμα της Βουλγαρίας μπορεί να έχει περαιτέρω Προεκτάσει και επιπτώσει. Όσον αφορά τώρα τι πληροφορίε που μας έχουν δώσει οι αρχέ ε, τη ε, Βουλγαρία, ε, οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν στο τέλο του καλοκαιριού. Το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων θα το χρησιμοποιήσει η Eurostat στο πλαίσιο των επισκέψεων που όπως σας είπα θα ακολουθήσουν στη Βουλγαρία. Όσον αφορά την ταχύτητα αναθεώρησης του αναθεωρημένου κανονισμού που εκχωρεί ενισχυμένες αρμοδιότητες στη Eurostat, η Eurostat ε, θα χρησιμοποιήσει τις διευρυμένες αρμοδιότητές της στο πλαίσιο των εργασιών που διεξάγει. Κυρίες και κύριοι λοιπόν, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την προσοχή σας και κυρίω θέλω να ευχαριστήσω για την ευρεία και αμέριστη υποστήριξη προς την πρότασή μας που είναι η πρώτη νομοθετική πρόταση της δεύτερης Επιτροπής Μπαρόζο. Η έγκριση λοιπόν της πρότασης αυτής είναι εκ των όνου κάνευ για να έχουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα οικονομική και νομισματική ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε και για την γενοδορία σας απέναντί μας που πρέπει να πω ότι πράγματι εμείς δεν επιδείξαμε τη δέουσα προσοχή ε, σε αυτά που λέγατε. Λυπάμαι πάρα πολύ που ε, υπήρξαν αυτά τα χειροκροτήματα και η φασαρία που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά που ελέγονται. Σε αυτό λοιπόν το σημείο Θέλω να πω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Οι ε, ψηφοφορίες ε, θα λάβουν χώρα για το θέμα αυτό την Πέμπτη το πρωί. Ε, θα διακόψουμε για δύο λεπτά τη συνεδρίασή μας και μετά θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας για να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. say something? E, Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Καθίστε.